Kolleginnen um Σας ζητώ συγγνώμη αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχα ωστόσο μια ε, ομάδα νεαρών ε, βουλευτών, οι οποίοι, νεαρών Πολωνών βουλευτών που ήταν ε, μαζί μου στο γραφείο μου και μιλήσαμε, ίσως Ουκρανών υποπρόεδρος, για τις εξελίξεις στο Μίνσκ Ουκρανών. Μάλιστα και εγώ ίδιος επισκέφθηκα το Κίεβο, το ε, Σαββατοκύριακο μίλησα με τον πρόεδρο εκεί. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις στην χώρα τους και ταυτόχρονα να διεξάγουν πόλεμο. Έχουν δηλαδή εμπόλεμη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά προχωρεί η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Μόλις τώρα τα συζήτησα βέβαια αυτά μαζί τους. Δεν θα τα συζητήσουμε τώρα. Αλλά για μας αυτό που συνέβη σήμερα με την κυρία Σαφτσένκο είναι απολύτως απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την απόφαση διότι βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα και σε καμία δικαιική βάση. Αν συμφωνείτε λοιπόν να μου επιτρέψετε να εγείρουμε διαμαρτυρίες ε, εκ μέρου σα δηλαδή, όπως άλλωστε προτίθεται και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι κανεί δεν ενίσταται εξ ημών, άρα έτσι θα κάνουμε. Ενστάσεις για την ημερησία διάταξη. Όχι. Τις ανακοινώσεις τις έκανα. Άρα προχωρώ τώρα στην συνομιλία με την κυρία Τσάτσεβα, πρόεδρο της Βουλγαρικής Βουλής, και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της ε, νοτιοανατολικής, διαδικασία, νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Συνεργασίας. Πολύ χαίρομαι που προσήλθατε σήμερα ενώπιον μας, κυρία Πρόεδρε. Ήδη συζητήσαμε και μαζί σας και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως και με τον ΟΟΣΑ μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτής της οργανώσεως της οποίας ηγείστε να ενταθεί η συνεργασία και ιδίω συνεργασία σε τομείς δημοκρατίας και ανάπτυξης θεσμών. Νομίζω ότι όλοι εκεί συμβάλλουν, όλες οι πλευρές συμβάλλουν με τον τρόπο τους, αλλά δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία και συντονισμός. Και για χώρες όπου με τον τρόπο αυτό, με τη συνεργασία και τον συντονισμό θα επιτύχουμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας και ίσως θα πρέπει να οργανώσουμε κοινή συνάντηση προ των θερινών διακοπών μαζί με τους προέδρους της Συνοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΩΣΑ και εσάς βεβαίως. Ευχαριστώ και πάλι που λάβατε τον κόπο να προσέλθετε ενώπιον μας. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι και από τα κοινοβούλια των κρατών μελών που βρίσκεστε εδώ, και μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, της Διακοινοβουλευτικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που μας δίδετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε πνεύμα συνεργασίας Είναι ένα εξαιρετικό φόρουμ η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μιλήσαμε, ξεκινήσαμε με πολιτικά θέματα και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα πάρα πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζεται ε, στα πλαίσια της ε, μεταναστευτικής κρίσης, λέει ο Μιλήτρια. Οι χώρες της περιοχής από μόνες τους δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις οι οποίες είναι μπροστά τους. Δεν έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις κρίσεις αυτές. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες εκκλήσεις για απομονωτισμό και εσωστρέφεια είναι κάτι το οποίο ακούγεται όλο και περισσότερο. Εγώ λοιπόν συμμερίζομαι τις απόψεις των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων της Ευρώπης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την ευρωπαϊκή συνεργασία και για την Ανατολική Ευρώπη. Οι κίνδυνοι που έχουμε μπροστά μας είναι κοινοί. Οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις λόγω ακριβώς των πάρα πολλών αλλαγών που συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και ακόμα και στη Μαύρη Θάλασσα. Και γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος εδώ από την έλλειψη κοινής αντίληψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ε, με τις προκλήσεις, αλλά θα ήθελα να σταθώ και σε κάποια θετικά στοιχεία της περιοχής. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση λοιπόν της Νοτιοανατολικής Συνεργασίας δημιουργήθηκε εδώ και 20 χρόνια. Στο Βουκουρέστι λοιπόν ξεκινήσαμε σε μια επίσημη βάση συνεργασίας υιοθετώντας ε, την ιδρυτική μας διακήρυξη όπως επίσης και τον κανονισμό με βάση τον οποίο εργαζόμεθα. Έχουμε θεσμικοποιήσει περαιτέρω την ε, κοινοβουλευτική μας συνεργασία. Έχει γίνει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για μας και θα θέλαμε να καταστήσουμε και τις σχέσεις μας με τα ευρωπαϊκά όργανα ε, πιο αποτελεσματικές σε θεσμικό επίπεδο, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιας και είμαστε και εμείς φύση φύσεως σώμα. Γεωγραφικά μιλώντας, η περιοχή την οποία εκπροσωπούμε περιλαμβάνει χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι ήδη κράτη-μέλη. Κάποιες άλλες χώρες είναι υποψήφιες ε, δυνητικά χώρες και υπάρχει και άλλη μια ομάδα επίσης χωρών οι οποίες ονομάζονται όπως γνωρίζετε ε, χώρες διεύρυνσης, είναι στη φάση της διαδικασίας για τη διεύρυνση. Έτσι ώστε λοιπόν θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και να βασιστούμε και στο υδροτικό μας έγγραφο, στο καταστατικό μας έγγραφο και με αυτή τη βάση σας ευχαριστούμε γιατί ε, επιτρέπετε και εσείς με τις ενέργειές σας να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για το μέλλον, να ανταλλάξουμε βέλτιστες, τις βέλτιστες πρακτικές και να σταθούμε πιο αποτελεσματικοί. Σήμερα ε, θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην κατάσταση της περιοχής. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αν η συνεργασία μας σε θεσμικό επίπεδο καταστεί αποτελεσματικότερη νομίζω ότι θα προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως και τα κοινοβούλια των κρατών μελών που συμμετέχουν στην διακοινοβουλευτική αυτή μορφή συνεργασίας, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επαναλάβω ότι εμείς δεν έχουμε διαφορές σε σημαντικά θέματα, όπως οι πολιτικές και τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την ενίσχυση των μορφών συνεργασία μας. Η υπογραφή ενός εγγράφου ανεξαρτήτως του τίτλου του εγγράφου αυτού δεν είναι κάτι το οποίο αφέ αυτού έχει σημασία. Ένα τέτοιο έγγραφο που θεσμοποιεί τις συνεργασίες μας θα πρέπει να εδράζεται σε κοινές πολιτικές αντιλήψεις έτσι θα ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε θεσμικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Η αντιπροσωπεία σήμερα εκπροσωπείται από Έλληνες, ε, Βοσνίους, ε, Μολδαβούς και επίσης ε, κοινοβουλευτικούς από το Κωσυφοπαίδιο. Ε, στη Σερβία και στην Μακεδονία λέει η ομιλήτρια ε, διεξάγεται προεκλογική εκστρατεία οπότε ε, δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στις συζητήσεις. Νομίζω όμως ότι και αυτοί επιθυμούν τη στενότερη συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στη δική μας συνέλευση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προεδρεύουσα λοιπόν του συγκεκριμένου οργάνου να μου επιτρέψετε να σας περιγράψω το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, κινούνται οι εργασίες μας ε, και η συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει σήμερα. Να υπογραμμίσω λοιπόν τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πίεση στην περιοχή είναι μια σοβαρότατη απειλή για τη σταθερότητά της όλοι οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων στις συζητήσεις τις οποίες είχαμε σήμερα το πρωί συγκέντρωσαν την προσοχή τους στην ανάγκη η οποία υπάρχει για να δημιουργηθούν κοινέ ε, ε, αντιλήψεις για την επίλυση του θέματος αυτού. Ε, θα πρέπει φυσικά να σεβαστούμε και τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία που το υπογραμμίζουμε αυτό. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία για τις, χώρε για τις χώρες της περιοχής να αποκτήσουν ε, πλήρη έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, να τηρήσουν τις ανηλυμένες τους υποχρεώσεις και να εφαρμόσουν όλες επαναλαμβάνω οι χώρες της περιοχής της υπογραφή σε συμφωνίες στο παρελθόν στον τομέα της ε, επανεισδοχής. Η συμφωνία η οποία υπεγράφει ε, την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία ήταν απαραίτητη. Από εδώ και πέρα πρέπει να διανύσουμε έναν δρόμο ιδιαίτερα μακρύ για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα υπεσχημένα και να σεβαστούμε και τις εθνικές νομικές ρυθμίσεις αλλά και το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι η δημιουργία μιας πραγματικής μεταναστευτικής πολιτικής κοινή για τα ευρωπαϊκά όργανα είναι μια θα έλεγα αναπόφευκτη διαδικασία αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Είμαστε ένα περιφερειακό και πρέπει να καταστούμε ένα σημαντικό περιφερειακό φόρουμ λοιπόν και ως προς την κατεύθυνση αυτή να σας παρουσιάσω κάποιες προτεραιότητες σημαντικές όχι μόνο για την Βουλγαρική Προεδρία αλλά για το σύνολο της διακοινοβουλευτικής μας συνελεύσεως. Θα πρέπει να υπάρξουν διασυνδέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες χώρες στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών αλλά και ενέργειας. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Όταν υιοθετούμε σε εθνικό επίπεδο μέτρα στον τομέα αυτό δεν θα πρέπει να είναι ε, ε, θα έλεγα ε, κάτι το τυχαίο αλλά θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ενισχύεται η διασυνοριακή συνεργασία, να αυξάνεται η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων. Οι οικονομίες μας είναι όλο και πιο συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Τα θέματα αυτά τα έχουμε ήδη συζητήσει αρκετά αναλυτικά. Έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν αρκετά ψηφίσματα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νομική πράξη που έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα προβλήματα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Έτσι θα ενισχύσουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα και θα ενισχύσουμε και την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Η διαφοροποίηση προμήθειας είναι σημαντικό πρόβλημα και το υπογραμμίζουμε ιδιαίτερως. Να συγκεντρώσω τώρα την προσοχή μου σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ανάγκη που υπάρχει ε, και την ευκαιρία που έχουμε σαν διακοινοβουλευτική συνέλευση της συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να καταστούμε πρωτοπόρος οδηγός στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των χωρών αυτών. Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν ε, αναλάβει την υποχρέωση να επιδιώξουν την ευρωπαϊκή προοπτική. Όπως προείπα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ένταξης στην διαδικασία αυτή Κάποιες χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τις χώρες υποένταξη ή τις χώρες που είναι στην προετοιμασία της διαδικασίας ένταξης. Απαιτείται στενότερη συνεργασία και περισσότερες προσπάθειες και από πλευράς της δικής μας διακοινοβουλευτικής συνέλευσης αλλά και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαι πεπισμένη ότι εφόσον συνεργαστούμε περισσότερο και στενότερα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια ισότιμη εταιρική σχέση. Η βουλγαρική αντιπροσωπεία πρότεινε τον προηγούμενο μήνα να γίνει μια πρόταση για μια κοινή συμφωνία τι σημαίνει μια κοινή συμφωνία η οποία να βασίζεται στους κανόνες τους διαδικαστικούς τους οποίους εφαρμόζουμε. Ανεξάρτητα λοιπόν από τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα ονοματίσουμε τη συγκεκριμένο έγγραφο, αν θα είναι μνημόνιο κατανόησης ή συμφωνία συνεργασίας, το έγγραφο αυτό θα πρέπει να καθορίζει με σαφή τρόπο τις πολιτικές τις οποίες θα πρέπει από κοινού να επιδιώξουμε, όπως επίσης και να κατά κάποιο τρόπο να σταθεροποιήσουμε τις μορφές συνεργασίας μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπρόκο για την θετική απάντηση στην επιστολή την οποία έστειλα πριν μερικούς μήνες ήταν ένα πρώτο βήμα το οποίο είχε σαν στόχο την αποκατάσταση της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο όργανα μας. Ακολουθούμε διαφορετικές πορείες προς το παρόν σε επίπεδο διαδικασίας αλλά μπορούμε με κοινέ συναντήσεις να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας αυτή. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον βήμα προς τα εμπρό το οποίο θα βελτιώσει την εικόνα της διευρωπαϊκής συνεργασίας αυτής. Εφόσον καταφέρουμε λοιπόν στο μέλλον και με τη βοήθεια την δική σας και των εμπειρογνωμόνων και της εμπειρογνωμοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσουμε και την θεσμική μας συνεργασία η οποία θα είναι απαραίτητη και ευεργετική για όλες τις χώρες της περιοχής και κυρίως για όλους τους πολίτες της περιοχής στην αρχή της εισαγωγής μου υπογράμισα την ανησυχία μου για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε συγκυριακά. Θα ήθελα να κλείσω με μια πιο αισιόδοξη διαδήλωση. Όλα τα μέλη και από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη διακοινοβουλευτική μας συνέλευση θεωρούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την ευρωπαϊκή προοπτική, στην ευρωπαϊκή καλύτερα προοπτική. Περιμένουμε λοιπόν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, από να συνενέσουν στην αποδοχή των κοινών αυτών προσπαθειών και επαναλαμβάνω αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες των χωρών και τις χώρες οι οποίες είναι στην, σε επίπεδο ε, προόδου προς την διαδικασία ένταξης η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μας θα μας καταστήσει ικανούς να βελτιώσουμε την κυριαρχία του κράτους δικαίου, την ε, απόλυτη και πλήρη εφαρμογή των δημοκρατικών αξιών στις χώρες μας και φυσικά να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη απαιτείται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις χώρες της περιοχής. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την δυνατότητα αυτής της ανταλλαγής απόψεων. ο πρόεδρος Έλμαρ Βρόκ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ανάπτυξη των θεμάτων σας, για το μήνυμα που δώσατε και πρώτα δίνω τον λόγο στον κύριο Κόβατσεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάτσεβα. Καλώς ήρθατε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά σας της προεδρευούσης της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σωστά είπατε ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία έχει εξαιρετική σημασία. Έχει επίσης μεγάλη σημασία η ανταλλαγή καλών πρακτικών για να βελτιωθεί η κοινοβουλευτική, η εποπτεία. Και μάλιστα σημαντικά. Η συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σημαντική διότι βοηθεί τις χώρες της περιοχής να υπερβούν ελλείμματα, ελλείψεις που έχουν από το παρελθόν, ελλείψεις που έχουν από το παρελθόν. Και για την ώρα είναι το ο μόνος μηχανισμός ενίσχυσης της συνεργασίας που διαθέτουμε. Όλα όσα αναφέρατε για την σύναψη συμφωνίας ή μνημονίου συμφωνίας με, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά απηχούν και τους βασικούς μας στόχους. Ωστόσο, Θα ήθελα με την ευκαιρία να θέσω μια ερώτηση που ίσως σας φανεί κάπως έμεση. Με ενδιαφέρει η συνεργασία και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, διότι όλες αυτές οι χώρες οι οποίες ακολουθούν την οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένταξη και θέλουν να συνεργαστούν, θα πρέπει να υπερβούν τα τεράστια κολλήματα που απορρέουν από τις διαφορές μεταξύ τους στον ψηφιακό τομέα για παράδειγμα όταν χρειαστεί να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της περιοχής καλείστε να κατεβάλλετε τεράστια τέλη περιαγωγής θα ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω έκκληση, να απευθύνω έκκληση σε όλες τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αρχίσουν ήδη από τώρα να υιοθετούν κάποια από τα νομοθετήματα που διέπουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Γνωρίζω ότι οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών ίσως να σταθούν αντίθετες. Είναι όμως πολύ σημαντικό αυτό για την ένταση της συνεργασίας στην Επιτροπή και θα σημάνει και ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, διότι αυτά είναι εμπόδια στη συνεργασία. Θα ήθελα εξάλλου να εκφράσω και μια ευχή για επιτυχία της ε, προσπάθειάς σας και ασφαλώς μπορείτε να βασίζεστε και στη δική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Πρόκ, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κυρία Τσάτσεβα. Είμαι και πρώην εισηγητής για την χώρα σας, την Βουλγαρία. Σας καλωσορίζω λοιπόν και με την ιδιότητα αυτή. Βλέπω ότι τα 13 μέλη της οργανώσεώς σας, της, της ε, συνελεύσεώς σας, 7 από ε, τις χώρες αυτές δεν είναι μέλη της Ένωσης για την ώρα έχετε τον αξιέπαινο στόχο να ενισχύσετε τις γειτονικές σχέσεις, τη συνεργασία, αλλά μοιράζεστε και πολλά και επίμονα προβλήματα. Ορισμένα τα έχουμε συζητήσει προημερών ε, στην παρούσα Επιτροπή Εξωτερικών όταν συζητήσαμε τους μηχανισμούς επαλήθευσης και την εφαρμογή τους στην Βουλγαρία και Ρουμανία για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το οργανωμένο έγκλημα, η αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης και άλλα σχετικά. Όντως λοιπόν αντιμετωπίζεται κάποια θεμελιώδη κοινά προβλήματα. Ασφάλεια προμήθειας ενέργειας, η εξάρτηση πολλών από τις χώρες της περιοχής, από ένα βασικό, ένα μείζωνα προμηθευτή φυσικού αερίου. Επίσης, πηγές εμπορίου, παράνομου εμπορίου όπλων θα τις βρείτε συχνά σε κάποιες από τις χώρες σας. Παράνομος οπλισμός, ο οποίος καταλήγει στην Δυτική Ευρώπη. Και αυτό το οποίο θίξατε εσείς, δηλαδή το προσφυγικό, που είναι η μεγαλύτερη κρίση που πλήττει την Ευρώπη. Και ιδίω το τμήμα εκείνο της Ευρώπης που εκπροσωπείτε εσείς εδώ. Διερωτώ με σε ποιο βαθμό θα μπορέσετε να συμφωνήσετε μεταξύ σας για τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει να ξεπεραστεί το μέγα αυτό πρόβλημα. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το, μάλλον το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο σας βοηθεί ή ενδεχομένως όχι την επίλυση αυτής της κρίσης. Ε, υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να αναθεωρηθούν ή και να παραξεταστούν ή και να αναθεωρηθούν ενδεχομένω η λειτουργία της συνθήκης για τους πρόσφυγες ή και της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις οποίες βασίζονται τα δικαιώματα πολλών από τους ανθρώπους που προσέρχονται στην Ευρώπη ως πρόσφυγες ή και ως μετανάστες. Μεγάλη αριθμή από τα πρόσωπα αυτά έρχονται από δύο χώρες που συμμετέχουν στην ε, συνέλευσή σας, δηλαδή από το Κόσοβο και την Αλβανία. 70.000 από το Κόσοβο, 60.000 από την Αλβανία. Άρα, σημειώνονται κάποια πραγματικά προβλήματα και διορωτώ εάν θεωρείτε ότι διαθέτει τους μηχανισμούς για να τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος, δεν ακούμε δυστυχώς το όνομα που εκφωνεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Πολύ χαίρομαι που μπορώ εδώ να συμμετάσχω και εγώ στην συνάντηση αυτή και να σας μιλήσουμε για την διαδικασία για τη συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες και οι συζητήσεις που έχουμε εδώ θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε το όργανο αυτό να αποτελέσει μια πλατφόρμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής σε όλα τα επίπεδα. Και στη συνέχεια συνεργασία βέβαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θεσμική συνεργασία ανάμεσα την δικιά μας κοινοβουλευτική συνέλευση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να μπούμε και στον δρόμο που θα μας οδηγήσει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα βοηθήσει την ολοκλήρωση τη θεσμική στην περιοχή. Θα μας βοηθήσει επίσης να εναρμονίσουμε και την ομοθεσία να ισχύσει και σε εμά το κοινοτικό κεκτημένο. Τώρα, ε, να δούμε για τα θέματα της ε, ατζέντα της Μολδαβίας. Υπάρχουν κάποια θέματα προτερότητα για τις μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις ε, επιθυμίες, τις προπτικές που βλέπουν οι πολίτες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου εξωτερικών υποθέσεων. Τα προβληματικά ζητήματα, οι προβληματικοί τομείς είναι ίδιοι και είναι ακριβώς αυτοί για τους οποίους η κυβέρνηση έθεσε προτεραιότητες. Χρειάζονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις και πρέπει να ξεκινήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα που έγιναν στο παρελθόν. Το Κοινοβούλιο λοιπόν και η κυβέρνηση εξακολουθούν να θέλουν την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και η συνεργασία βάσει αυτής της ε, συμφωνίας θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές μας στο δομέα της ενέργειας, στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει επίσης να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες μας και να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής τους. Θα μας βοηθήσει επίσης να μειώσουμε τις κρίσεις και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στην παγίωση της δημοκρατίας, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακόμα κάτι πολύ σημαντικό θα ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί των χωρών μελών. Τώρα πιο συγκεκριμένα για τη Μολδαβία σας διαβεβαιώ ότι το σημερινό κοινοβούλιο και η σημερινή κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν κάθε ευκαιρία συνεργασίας που παρουσιάζεται και προκειμένου να επωφεληθούμε από οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προκειμένου όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να επωφεληθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη στήριξή σας, για τη στήριξη που προσφέρετε στη χώρα μου. Και είμαι σίγουρη ότι η πλατφόρμα αυτή συνεργασίας της Ανατολικής Ευρώπης θα είναι επωφελής τόσο για την ίδια την κοινοβουλευτική συνέλευση, όσο και για τους πολίτες των χωρών που συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. <laughs> Ähm, ε, ευχαριστώ, θα μιλήσω ρουμανικά. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα περάσω στην ουσία. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κρίση εκείνη των προσφύγων και του μεταναστευτικού. Το 2009 με έκθεση για τη Eurodac λέγαμε ότι η καλύτερη νομοθεσία μπορεί να βελτιώσει όλα τα συστήματα και ότι συγχρόνως μπορούν να λυθούν όλα τα σοβαρά προβλήματα που έχουν οι χώρες οι οποίες έχουν πολλούς παράνομους μετανάστες. Αυτά το 2009. Έκτοτε τα πράγματα έχουν προχωρήσει και πρέπει να αντιδράσουμε έντονα νομοθετικά. Ο κύριος Βανόρντεν είχε δίκιο. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, ακόμα και η κοινοτική νομοθεσία. Και θα σας κάνω μία συγκεκριμένη πρόταση. Τη σήμερα ημέρα για το πολιτικό άσυλο Για να θεωρηθεί δηλαδή κάποιος πρόσφυγας, που αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση, όχι σε προσωρινή, όπως είναι ο πόλεμος της Συρίας, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή προστασία. Προσωρινή προστασία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό το σωστό. Το σωστό θα ήταν οι χώρες να προσφέρουν πρώτον προσωρινή προστασία και στη συνέχεια να εξετάσουν κάθε περίπτωση χωριστά και μετά να προσφέρουν την μόνιμη προστασία που σίγουρα πολλοί χρειάζονται. Αυτό θα ήταν μια τροποποίηση της νομοθεσίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αντιδράσει και πολύ γρήγορα να ληφθεί σχετική απόφαση. Η κυρία Τσάτσεβα από τη Βουλγαρία ε, μας το είπε ότι στη Βουλγαρία προσπαθούν να τροποποιήσουν την νομοθεσία και εμείς στη Ρουμανία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ο πρόεδρος Γιωχάνης ανακοίνωσε ε, τροποποίηση της νομοθεσίας προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Γιατί η ιδέα εδώ είναι να δώσουμε ευκαιρία για να υπάρξει μία δίκαια, μία σωστή λύση. Είναι σωστό να δώσουμε προστασία σε κάποιον που την χρειάζεται, αλλά δεν είναι σωστό να προσφέρουμε προστασία σε κάποιον ο οποίος μπορεί να δώσει ψεύτικες πληροφορίες. Λάθος. Δεν γενικεύω αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Πρέπει να αντιδράσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτό. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχει μικρόφωνο αναμένο ο πρόεδρος Μπρόκ. τη σημερινή συνάντηση του ΣΥΣΠΑ και της ΑΦΕΤ ως την αρχή μιας ε, επικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάγια θέση μας είναι ότι η υποστήριξη της ένταξης των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα την υποστηρίζαμε, αλλά πάντα με βάση την αρχή της αιρεσιμότητας. Η Ευρώπη διέρχεται σήμερα μια πολυεπίπεδη ιστορική κρίση, οικονομική, προσφυγική, μεταναστευτική, τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει μπροστά της δύο εναλλακτικές λύσεις. Ή να υπερασπίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου ή τη λογική των κλειστών θυρών και του εθνικού απομονωτισμού. Η προσφυγική κρίση υπερβαίνει την ατομική δυνατότητα των χωρών και ως εκ τούτου πρέπει να τύχει συλλογικής και συντονισμένης αντιμετώπισης. Είτε θα διαμορφώσουμε μια κοινή πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης ή η κρίση θα μας καταπνίξει, θέτοντας και θέμα επιβίωσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μονομερείς ενέργειες και το κλείσιμο των συνόρων δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, έπληξαν άμεσα την πατρίδα μου την Ελλάδα με τον εγκλωβισμό μεγάλου αριθμού προσφύγων. Θεωρούμε θετικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εργαστούμε σκληρά και γρήγορα για την υλοποίησή της. Και το υπογραμμίζω αυτό γιατί ενώ από το Σεπτέμβρη υπήρχε απόφαση για τη μετεγκατάσταση από τις χώρες πρώτης υποδοχής 160.000 προσφύγων προς, τις, τα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής εγκρίθηκαν μόν, μόλις 2.000 και πραγματοποιήθηκαν 584. Τελειώνοντας, τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων απαιτεί άμεση εφαρμογή όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν για τη μείωση των ροών. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του στόχου της φύλαξης των συνόρων και του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου για το άσυλο. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων συνόρων μας, καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φύλαξης Συνόρων και Αχτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέτοια μέτρα τα έχει προτείνει το Κοινοβούλιο ήδη από 15 ετίας. Βέβαια, Κομισιόν και Συμβούλιο Υπουργών έρχονται πάντα με μια καθυστέρηση. Ο κ. Καβούζογλου τώρα από την Τουρκία. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η συμφωνία αυτή ελπίζω να ανοίξει προοπτικές και να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυτό το οποίο επιθυμεί είναι την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσω πολιτικών οι οποίες να είναι συμβατές με τις πολιτικές της Ευρώπης. Η κρίση των μεταναστών έχει δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα, δεν θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα άλλο χώμα, σε ένα άλλο θέμα, Όπως είπα τα μέλη μας είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες στην διαδικασία ένταξης, οι χώρες που οδεύουν προς την διαδικασία ένταξης. Για να προχωρήσουν τα πράγματα χωρίς δυσκολίες θα πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω πολιτικές συγκρούσεις, θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να κατοχυρωθεί σαν στόχος, να διασφαλιστεί η ε, διακίνηση ελεύθερη των πολιτών των χωρών που το επιθυμούν. Ευχαριστώ ο Κούκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την τοποθέτηση της Προέδρου της Νότιο-Ανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Είναι όντως σημαντική η συνεργασία με τα κοινοβούλια των χωρών της περιοχής. Αντιμετωπίζουμε όλοι πολλές προκλήσεις και χρειαζόμαστε την κοινοβουλευτική συνεργασία και τον κοινοβουλευτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. γιατί η συνεργασία αυτή έχει και σημαντική επιρροή στην εφαρμογή των ιδεών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενταχθεί στον διάλογο αυτό. Θεωρούμε επίσης ότι για να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής συνεργασίας, αυτό θα βελτιώσει και την ποιότητα της διαδικασίας διευρύνσεως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε διαρκή διακοινοβουλευτικό διάλογο με τις χώρες της περιοχής. Οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές από τις περισσότερες από τις χώρες της ε, νοτιοανατολικής συνεργασίας συμμετέχουν τακτικά στις συναντήσεις αυτές. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ιδέα μιας ενδεχόμενης στενότερης συνεργασίας με τις χώρες της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής συνεργασίας, αλλά αντί για τυποποιημένες σχέσεις, εγώ θα συνιστούσα να συνεχίσουμε με πιο εύκαμπτες μορφές συνεργασίας. Για παράδειγμα, τακτικό διάλογο για επίκαιρα θέματα της ε, διευρύνσεως συμμετοχή των Ευρωβουλευτών σε συναντήσεις βουλευτών της Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και πάνω και άλλες σχετικές ευκαιρίες, διότι αυτή η συνεργασία εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα όλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μπρόκ, αλλά δυστυχώ χωρί μικρόφωνο, ό,τι ακούμε από άλλα μικρόφωνα. Εσεί ευχαριστώ κύριε Μπρόκ, θα συνεχίσω όμω στα αγγλικά, διότι δεν υπάρχει μετάφραση από την αλβανική. Θα ήθελα πρώτα να πω Ρουμανία, μετά η Βουλγαρία. Έχουν τώρα την ε, Προεδρία της ε, Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας από πέρασε και τη δική μου χώρα. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία σε πολλού τομεί, ασφάλεια και αλλού. Εκτιμούμε πολύ το γεγονό ότι μα προσκαλείτε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών τη Ευρωβουλή για να συζητήσουμε περί ενισχυμένη συνεργασία. Διεξάγουμε συζήτηση και μεταξύ μα πού δηλαδή θα έχει την έδρα τη η διαρκή γραμματεία. Μέχρι ότου λυθεί το πρόβλημα, ίσω θα έχουμε ταχθεί όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι πιο εύκολο τότε γιατί θα έχουμε τι Βρυξέλλε ω έδρα τη Διαρκικού Γραμματεία. Τέλο πάντων, μέχρι τότε θα ίσω πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Οφείλω να πω λίγα λόγια για το βασικό θέμα που συζητείτε και εσεί εδώ, το προσφυγικό. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την Τουρκία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, που συνήψαν τόσο σημαντική συμφωνία την προηγούμενη Πέμπτη η οποία μπορεί να αποτελέσει το σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Όπως συζητήθηκε όμως την προηγουμένη Πέμπτη, και στις ευχαριστίες που δόθηκαν στην Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ως ευχαριστία δίνεται ας πούμε και η αναθεώρηση του συστήματος προξενικών θεωρήσεων Νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλων των αντιπροσωπιών της ανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων και για ε, πολίτες του Κωσόβου. Αυτό θα είναι καλό, διότι θα αντιμετωπίσει έτσι και τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής Βαν Όρντεν. Ε, πέρσι, αυξημένος αριθμός Αλβανών από το Κόσοβο ζήτησαν άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του φετινού χρόνου λόγω της, ή στην καλή συνεργασία Αλβανίας, Κόσοβου και ευρωπαϊκών χωρών μελών. Συμπεραίνοντας λοιπόν, είναι σωστό να επανεξεταστεί το, το δυνατόν συντομότερο η διευκόλυνση για προξενικές θεωρήσεις για το Κόσοβο. Ο Πρόεδρος. Δεν ακούμε τη δυστυχώ. Εσείς έχετε το λόγο, σας ευχαριστώ. Ε, ε σας ευχαριστώ και Μπροκ. Πρόεδρε. Και Προεδρεύουσα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Διδικασίας για τη Συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε δυνατότητε συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση για την Νοτιοανατολική Συνεργασία. Το 1996 συμμετείχα στην αρχή της συνεργασίας αυτής. Είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που ξεκίνησε από το Σύμφωνο Σταθερότητας για την περιοχή. Εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να δούμε ό,τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, οι χώρες αυτές βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ένταξης. Άλλες είναι οι άλλες περιμένουν να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις κλπ. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική συνεργασία πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κλειδί για αυτές τις χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως όταν αναφερόμαστε στις επιτροπές των κοινοβουλίων των χωρών αυτών για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ένα πρόβλημα που το ακούσαμε ήδη είναι εκείνο το ότι Το έχουμε ακούσει από πολλούς μέχρι τώρα. Είναι το θέμα του προσφυγικού που έχει να κάνει με τη γεωγραφική βέβαια θέση των χωρών αυτών. Πρέπει να τηρούνται οι ευρωπαϊκές αρχές, να σεβόμαστε την συνθήκη Σέγγεν, τις διάφορες διμερείς συμφωνίες και βεβαίως να προσφέρουμε προστασία σε εκείνους τον οποίων η ζωή κινδυνεύει. Πρέπει να σεβόμαστε τις ευρωπαϊκές αξίες και σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την κοινοβουλευτική συνεργασία για να ενισχύσουμε και τις οικονομικές μας σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων χωρών στην περιοχή. Το γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχουν ακραμούντα ζητήματα μεταξύ των χωρών μελών της αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτική αυτής συνέλευσης. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε διάλογο κάθε φορά που αυτό χρειάζεται και ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε τις νοτιοντολικές ε, χώρες της Ευρώπης στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραμείνει βέβαια μια προτεραιότητα. Σήμερα, αργότερα, θα συζητήσουμε για την Βοσνία Ριζεγοβίνη και θα συζητήσουμε και για την Αλβανία. Θα δείτε λοιπόν όταν φτάσουμε εκεί πώς ε, προχωράει η διαδικασία κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει, παρουσιάζει την έκθεσή της για την κατάσταση πρόοδου των χωρών αυτών και πώς αντιδράει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός ο μικροφόνο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αλβανικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να απευθύνω σε όλους σας χαιρετισμό. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω την Προεδρεύουσα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της διαδικασίας για τη συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα και πρέπει να σας πω ότι σέβομαι όλες τις απόψεις που ακούστηκαν. Ευθυγραμμίζονται, εξάλλου, με τις απόψεις και τις προσδοκίες των περισσότερων τουλάχιστον χωρών της περιοχής όσον αφορά την Ευρώπη. Όμως, θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα και αυτό είναι το κοσυφοπέδιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χώρες οι οποίες στήριξαν τη Συμφωνία Σταθερότητας με το κοσυφοπέδιο Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπερψήφισε τη συμφωνία αυτή. Θέλω επίσης δημόσια να κάνω έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνουν την κατάρχηση των θεωρήσεων για τους πολίτες του σκοσφοπεδίου. Βλέπετε, είμαστε η μόνη πια χώρα απομονωμένη στην Ευρώπη. Είμαστε η μόνη χώρα τις οποίες οι πολίτες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είμαστε η μόνη χώρα που δίνει δυνατότητες στους φοιτητές, στις επιχειρήσεις, οπότε Είμαστε η μόνη χώρα που βρίσκεται ακόμα σε απομόνωση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει συνεργασία με το κοσυφοπαίδιο και η οικονομία της χώρας ε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε πολλές περιπτώσεις η συμφωνία ΣΕΦΤΑ που έχει υπογραφεί με χώρες της περιοχής δεν εφαρμόζεται πλήρως. Τώρα, έρχομαι στο θέμα των 70.000 προσφύγων από το Κωσυφοπαίδιο. Το μέγεθος, το νούμερο, ναι, είναι τέτοιο. Από την άλλη μεριά γνωρίζω και την προηγούμενη κατάσταση όπου χώρες της Δυτικής ε, των Δυτικών Βαλκανίων, είτε πρόκειται για τη Μακεδονία, λέει ο μιλητή, είτε πρόκειται για το Μαυροβούνιο και για άλλου που έχουν δεχτεί ένα εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες. Συμφωνώ ότι η κατάσταση τότε ήταν διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Όμως το Κωσυφοπαίδιο υπάρχουν εγκληματικές συμμορίες που εποφελήθηκαν από την μετακίνηση αυτή από τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο και εγκληματικές αυτές οργανώσεις χρησιμοποίησαν δυνατότητες και διευκολύνθηκαν μάλιστα από τη μετακίνηση τόσων μεγάλων αριθμών Κωσοβάρων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι η κατάσταση στους θεσμούς του Κωσυφοπηδίου δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο Μερικές φορές μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας που παραβιάζεται. Αυτά έχω να πω όσον αφορά το θέμα των προσφύγων από το κοσυφοπέδιο, Αλλά η κατάσταση αυτή ίσχυε πριν από τρία χρόνια, το νούμερο δηλαδή των 70.000. Τώρα έχουν αυξηθεί κατά πολύ και δεν είναι δυνατόν Οι χώρες μέλη έχουν πολλές πληροφορίες από τους ίδιους τους Κωσοβάρους και πολλοί που μετακινήθηκαν επαναπατρίστηκαν, επέστρεψαν στο Κωσυφοπέδιο. Σίγουρα τα νούμερα έχουν αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα. Στηρίζω πάντως την πρωτοβουλία για την ένταξη όλων των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγχρόνως θέλω να σας πω ότι ο δημοκρατικός διάλογος που έχουμε για ειρήνη στα Βαλκάνια, κυρίως μεταξύ του Κωσυφοπεδίου και της Σερβίας, θα παραμείνει ευθύνη των αρχών του Κωσυφοπεδίου. Δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό. Σίγουρα και οι δύο πλευρές μπορούν να κάνουν πολλά. Παρά λοιπόν τα πολυάριθμα προβλήματα που υπάρχουν και στις δύο χώρες, ελπίζω ότι η πρωτοβουλία του CEPC e θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όλες οι χώρες μέλη της κοινοβουλευτικής αυτής συνέλευσης και με τις κοινέ τους προσπάθειες. Συγχρόνως ελπίζω οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτούν ότι η Ευρώπη είναι κοινό χώρος και όλοι πρέπει να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα σε αυτόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω όλους και να πω ότι αυτό το οποίο προέχει είναι να υπογραμμίσουμε κυρίως τη σημασία που έχουν συναντήσει σαν και αυτοί. Γιατί το λέω. Η σημασία, ε, το ρόλος μάλλον που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην υπόθεση αυτή πάρα πολύ σημαντικός. Η συνεργασία λοιπόν με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας ε, στην επίλυση της ε, κρίσης της μεταναστευτικής αν δεν ε, ολοκληρωθεί η συνεργασία με την Τουρκία δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές για την περιοχή μας και η οικονομία και το άσυλο και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική του ασύλου είναι θέματα στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλά μπορεί να κάνει, πρέπει να βοηθήσει τις χώρες αυτές ε, εντάσσοντάς τις στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Να βελτιώσουμε τις συνεργασίες μας και στα συγκεκριμένα θέματα, αυτά τα οποία συνδέονται με την μεταναστευτική κυρίως κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μπροκ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς αξιότιμοι βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Επιτρέψτε μου να πω πρώτα ότι η συζήτηση μου φάνηκε πολύ χρήσιμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συμμετασχόντες να ευχαριστήσω ιδίως τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών της Ευρωβουλής, τους εκπροσώπους και τις εκπροσώπους βέβαια της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Νότιο-Ανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, βλέπουμε ότι τα προβλήματα της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν και προβλήματα που συζητούνται και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας διαβεβαιώ και στρέφομαι προς εσάς ε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές ότι η σημερινή συζήτηση μας δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους και ελπίζω ότι η προσπάθειά μας, μας αυτή θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει στόχος που θα είναι δυνατός να επιτευχθεί για πολλές από τις χώρες της ε, περιοχής μας. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε εμείς να θεσπίσουμε τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την υπέρβαση της κρίσης του προσφυγικού. Πιστεύω ωστόσο ότι ίσως κληθούμε όντως να αναθεωρήσουμε κάποια στιγμή κάποιες από τις ισχύουσες συνθήκες. Θα χρειαστεί επίσης να σκεφτούμε σχετικά και με την ευρωπαϊκή και με τη διεθνή νομοθεσία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο παρελθόν και πώς θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του σήμερα. Έχουμε μεταφέρει στα εθνικά δίκαιά μας το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ένας εκ των συναδέλφων μας τόνισε και σωστά ότι τροποποιήσαμε τον νόμο μας για τη μετανάστευση και για τους ετουμένους άσυλο. Και είναι αληθές ότι και η Ρουμανική Βουλή ε, προτίθεται να πράξει κάτι παρόμοιο. Ωστόσο, ελπίζω ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην οργάνωσή μας, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετική φάση, σε διαφορετικό στάδιο της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένταξη, θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τις άλλες χώρες μέλη, θα πρέπει να συνεργαστούν και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής συνεργασίας και ασφαλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που με τις προσπάθειές τους επέτρεψαν την θεσμοποίηση των ε, διασυνδέσεων μεταξύ της κοινοβουλευτικής μας συνελεύσεως και του Ευρωκοινοβουλίου. Σας διαβεβαιώ θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει εμφολία ότι τα όσα πράττουμε σήμερα είναι χρήσιμα για όλες τις χώρες της περιοχής μας και βεβαίως ωφελούν τους πολίτες των χώρων μας. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Μπροκ για την ευκαιρία που μας δώσατε να προσέλθουμε σήμερα ενώπιόν σας, να συζητήσουμε μαζί σας, να θέσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν στις εργασίες της κοινοβουλευτικής μας συνελεύσεως της Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ με τη σειρά μου ειλικρινά και εγκάρδια, καθώς και και τους συναδέλφους της αντιπροσωπείας σας. Νομίζω ότι ακούστηκε από όλες τις τοποθετήσεις ότι θέλουμε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ και για το γεγονός ότι συζητήσατε όλα τα θέματα σήμερα που είναι σημαντικά για μας και ιδίω βέβαια το προσφυγικό. Επιτρέψτε μου να εκφράσω μια εντύπωση που έχω ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκαν καμιά φορά πλέον αλληλέγγυες από αυτές που ανήκουν και είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη αυτό από τον προηγούμενο χρόνο και ασφαλώς και το έχουμε σημειώσει εμείς αυτό. Και είναι και σωστό και σημαντικό να γίνει γνωστό. Και το θέμα αυτό του προσφυγικού που είναι πράγματι παγκόσμιο θέμα. Μιλούμε για 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή γύρω από το Ιράκ που ε, όμως ε, το βάρος το έχουν σηκώσει η Τουρκία, ο Λίβανος, η Ορδανία είναι μία από τις πηγές προσφύγων αυτών και αν εξετάσει κανείς τη γεωγραφική κατανομή και ειδικότερα τη χώρα σας ενδέχεται τώρα η χώρα σας να αποβεί νέος στόχος των διακινητών. Αυτά τα πράγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα δούμε να ανοίγονται και νέες οδοί από την Βόρεια Αφρική τώρα που έρχεται το καλοκαίρι σιγά σιγά και ησυχάζουν τα νερά των θάλασσών. Θα δούμε ήδη στα λιμάνια της Λιβύης που έχει αναλάβει πλέον το ρόλο των διακινητών το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις εκεί. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει η συνεργασία μας να παραμείνει στενή. Ήδη στην τελευταία διάσκεψη κορυφής η Μεγάλη Βρετανία έκανε σημαντικές προτάσεις για συνεργασία, το λέω αυτό προς την κατεύθυνση του Ευρωβουλευτού Βαν Όρντεν. Αντιλαμβάνεται και η Μεγάλη Βρετανία ότι δεν τα καταφέρνει και ούτε και η ίδια μόνη της να τα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και ότι αυτό αποτελεί και θεμέλιο για στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πολύ σύντομα θα είναι 60 εκατομμύρια πρόσφυγες και νομίζω ότι η αποκατάσταση της ειρήνης στην Εγγύς Ανατολή, το ξεπέρασμα των εγγενών προβλημάτων στην Αφρική, είναι ο τρόπος για να να αντιμετωπίσουμε στην ρίζα του το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον διάλογο και θα χαρώ πολύ να οδηγήσει σε πρακτικά συμπεράσματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στο περαιτέρω έργο σας. Kollegen, ist Fleckenstein? Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ο Φλέκενστάιν που είναι, ανάτος, ανάτος. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσουμε στο υπαριθμόν 4, έκθεση για την Αλβανία. Έχουμε κοντά μας τον εισηγητή μας κύριο Φλέκενστάιν. Νομίζω ότι η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο το πρωί, έτσι είναι. Αύριο το πρωί λοιπόν, ωραία. Και έχουμε και 163 τροπολογίες. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Φλάκενστάιν που έχει φτιάξει και 17 συμβαστικές τροπολογίες έχει ε, προβλέψει όλες τις σωστές λύσεις. Να κάνει την εισαγωγή τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε υπευλήθη το σχέδιο στις 17 Δευτέρου στην ΑΦΕΤ και συζητήθηκε μια πρώτη φορά. Από τον Ιούνιο του 2014 έχει το καθεστώς υποψήφιας χώρας η Αλβανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει σημαντικά βήματα πρόοδου σε πέντε τομείς προτεραιότητας για να μπορέσει να ανοίξει ή τέλος πάντων να εκδώσει τη σχετική σύσταση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Ιδίως για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που αποτελεί και προτεραιότητα για την αλβανική κυβέρνηση και φαίνεται πως και για το 90% του αλβανικού λαού η πιο σημαντική μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση δικαιοσύνης προβλέπεται να προχωρήσει γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες προτεραιότητες που είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστές. Η έκθεση βασίζεται στις πέντε προτεραιότητες και γι' αυτό δεν θα τα ξαναπώ, τα έχουμε συζητήσει ήδη και πέρσι. 163 τροπολογίες έχουν κατατεθεί, οι περισσότερες από τους κοιόδης εισηγητές βεβαίως, τους οποίους ευχαριστώ για την θετική και επικοδομητική συνεργασία. Υπήρξε υποστήριξη και για διάφορες συμβαστικές τροπολογίες για όλες τις θεματικές συμπληρώσει του κειμένου. Σε ένα σημείο δεν υπήρξε υποστήριξη εκ μέρου μου, όταν δηλαδή οι τροπολογίες τρέφονται ή τείνουν να ανατρέψουν το βασικό μήνυμα της εκθεσός μου. Δηλαδή τροπολογίες οι οποίες ζητούν για παράδειγμα να ανακοπεί εντελώς η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Το ίδιο και διότι δεν μου φάνηκε να διατηρείται επαρκώς η πολιτική ισορροπία τη εκθέσεως όταν δηλαδή έγιναν προσπάθειε προβολής ιδιαίτερα κάποιων συμφερόντων. Τα λέω αυτά διότι αυτά θα παίξουν, σημασία, θα παίξουν ρόλο συγγνώμη, και στην συζήτηση. βεβαίω και το θέμα τη προστασία των μειονοτήτων είναι σημαντικό. Όμω, αν αρχίσουμε τώρα να συζητούμε κάθε μειονότητα με παραγράφους ολόκληρες τότε νομίζω ότι θα διαραγούν τα όρια της εκθέσεως αλλά και της πραγματικότητας επιτόπου στην χώρα αυτή. Γι' αυτό και επιμέρους, σε επιμέρους θέματα βεβαίως διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις. Συνολικά λοιπόν έχουμε εκπονήσει 17 συμβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν τα πιο σημαντικά θέματα της εκθέσεως και της διαδικασίας μεταρρύθμισης στην Αλβανία. Ε, πρώτον επικοδομητικός πολιτικός διάλογος για τα θέματα ποινικοποίηση, για την αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης, για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την προστασία των μειωνοτικών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Εγκύψαμε και στην εργαδιοθήκη του ΟΣΑ και τον ρόλο που έπαιξαν στις τελευταίες εκλογές καθώς και στην τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας γενικότερα και στην πορεία προς την ένταξη, ε, το συζητήσαμε επίσης, την σημασία του επαγγελματικού πολυφωνικού δημόσιου ραδιοφώνου. Επίσης αυτό το συζητήσαμε και το θεωρούμε ως ένα στοιχείο κλειδί επίσης τις καλές γειτονικές διμερείς σχέσεις Αλβανίας αλλά και τον επικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας στην περιοχή ιδίως για την καταπολέμηση της Ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης και της ε, τρομοκρατίας. Εκεί επίσης αποδίδουμε μεγάλη σημασία. Κατόρθωσα εμείς και όλοι οι και εγώ προσωπικά να συμφωνήσουμε στις 17 ε, συμβαστικές τροφολογίες μέσα σε 30 μόλις λεπτά. Το εάν τώρα θα σημειωθεί κάποια διαφορά απόψεων σε ορισμένα σημεία, αυτό ενδέχεται να είναι αληθές. Ωστόσο θα φανεί καθαρά ότι έχουμε αρκετά ενία γνώμη για ε, τα θέματα αυτά και ότι φαίνεται καθαρά ότι η Αλβανία βρίσκεται στη σωστή πορεία. Παρόλο που θα θέλαμε κάποια πράγματα να γίνονται καλύτερα, σωστότερα ή και πιο γρήγορα. Πάντω η σωστή είναι η κατεύθυνση που λαμβάνουν οι Αλβανοί και χαιρόμαστε για την εξέλιξη αυτή. Ο Πρόεδρος, εσείς κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που προετοίμασε τις καλές συμβαστικές τροπολογίες και τον ευχαριστώ και για την καλή συνεργασία που είχαμε όταν ε, ετοιμάζαμε τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Έχουμε 17 λοιπόν συμβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν τα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα και βρίσκω πολύ συνενετικό και καλό τον τόνο της έκθεσης. Η έκθεση αυτή θα ήθελα να στηριχθεί ε, στην Αλβανία. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στη χώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει τους πολιτικούς της Αλβανίας να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Από τα πιο σημαντικά είναι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα είναι και αυτό που έχει συζητηθεί περισσότερο, αναφέρεται περισσότερο στην έκθεση και χαίρομαι που έχουμε καταλήξει σε κοινή γλώσσα από αυτού. Η Επιτροπή της Βενετίας τώρα ετοίμασε την έκθεσή της πριν από μερικές μέρες και ελπίζω ότι θα αποτελέσουν μια καλή κατευθυντήρια γραμμή για τις μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, χαίρομαι που πετύχαμε καλούς συμβιβασμούς για θέματα όπως είναι η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, την ε, ανάγκη να ακολουθήσει η χώρα της συστέασης του ΩΣΑ ή για θέματα εκλογικής διαδικασίας ή συνεργασίας στην περιοχή. Θέλω να υπογραμμίσω ένα ζήτημα με το οποίο έχω ένα μικρό πρόβλημα. Πρόκειται για τις τροπολογίες όσον αφορά την νομοθεσία, όσον αφορά την ε, νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ε, διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς πρόκειται για την νομοθεσία για το πώς αποφασίζεται ο διευθυντής του Συμβουλίου αυτού ραδιοφωνικών ε, σταθμών και αυτή η νομοθεσία είναι να αλλάξει και εγώ φοβάμαι ότι εδώ θα καταλήξουμε σε ένα θέμα ομοιρίας. Έχουμε κακή εμπειρία σε χώρες όπως είναι η Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Εγώ πρότεινα λοιπόν μια προφορική τροπολογία για τη συμβαστική τροπολογία 14. Και δύο άλλες προφορικές τροπολογίες πρότεινα που έχουν να κάνουν όμως με στοιχεία. Το ένα είναι για τον νόμο για την αποεγκληματοποίηση και η δεύτερη έχει να κάνει με το ρόλο των καταγγελόντων, των whistleblowers. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενη. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βάτματς. Να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον κύριο Φλέκενστάιν για τις προσπάθειες που έκανε για τη σύνταξη των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών για την έκθεση πρόοδου. Δεν θα ομιλήσω εκ μέρους του κύριου Γιούτσουκ, ο οποίος ήταν ο σκιώδης της ομάδας βέβαια, αλλά θα μεταφέρω κάποιες κοινέ απόψεις. Η Αλβανία λειτουργεί με επικοδομητικό τρόπο και έχει σταθερές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Έχουν υπάρξει σημαντικά βήματα πρόοδου για την επίτευξη των προγραμμάτων, των στόχων μάλλον, στον τομέα στον οποίο είχαν αναλυφθεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυφθεί μετά από υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθοριστικές για την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει βέβαια σήμερα η Αλβανία είναι πάρα πολλές και η κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά θετικά μέτρα για να τις αντιμετωπίσει συγκεντρώνει η αλβανική κυβέρνηση την προσοχή της σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας μηχανής και την κάθαρση της δικαιοσύνης. Συμπερασματικά, έχει σημασία να στηρίξουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην προσπάθεια εγγύηση των εθνοτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, των ευπαθών ομάδων και των Ρωμά. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φλέκενστάιν θα ήθελα να ομιλήσω εκ μέρους του Τάμας Μέσαριτς, σκιώδους ε, εισηγητή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεταξύ μας σήμερα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Φλέκενστάιν. Έχει προετοιμάσει μια καλή έκθεση, μια ισορροπή έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές. Οι περισσότερες από τις σκιώδεις τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνος και το σύνολο της έκθεσης θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Όπως είπε ο εισηγητής, η Αλβανία έχει κάνει αρκετά τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται, αν θέλετε, στο ότι έχει αποκτήσει ε, πρόσφατα σχετικά και την ιδιότητα της υποψηφίας χώρας. Μένει όμως να γίνουν ακόμα πολλά, έτσι ώστε να παραμείνει στην συγκεκριμένη πορεία που θα οδηγήσει στην ιδιότητα του μέλους. Σχετικά τώρα με τις συμβιβαστικές τροπολογίες, να αναφερθώ στην 16 για τις ασφαλείς χώρες. Η δική μας πολιτική ομάδα έχει κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τον κατάλογο. Συνήθως, αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση θα έλεγα μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα για τον κατάλογο των ασφαλών χωρών και γι' αυτό θα ήθελα το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας να διαγραφεί. Να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις ασφαλείς χώρες και στη δική μας Επιτροπή και στην Επιτροπή Λίμπε και μετά ίσως να συμπληρώσουμε τον κατάλογο. Υπάρχουν επίσης και συγκεκριμένες αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί. Βρίσκουμε ότι έπρεπε να υπάρξει αυτό. Επίσης γίνεται αναφορά και στην 134 η οποία έχει σχέση με την προστασία των υδάτων ε, ε, ενός συγκεκριμένου ποταμού στην Αλβανία. Ίσως ε, Βιώσα ακούσαμε ένα όνομα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξουν οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί το τίμημα και οικονομικό και περιβαλλοντικό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν τις τροπολογίες μας 137 και 138. Κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αναφερόμαστε στις πρόοδους που έχει σημειώσει η Αλβανία στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μάλιστα επισημαίνουμε τον επικοδομητικό ρόλο το οποίο διαδραματίζει στην περιοχή. Εγώ έχω εντελώ διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό. Δεν δημιουργεί συνθήκε καλή γειτονία με την Ελλάδα, με την οποία έχει προβλήματα όχι μόνο διότι καταπιέζει τα δικαιώματα τη ελληνική μειονότητα που υπάρχουν σε αυτή, έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη σε αυτό το θέμα, δεν θέλω να επεκταθώ. Έχει αναιρέσει η Αλβανία την υπογραφή τη σχετικά με τον καθορισμό τη ΑΟΣ των δύο χωρών και επιπλέον πρόσφατα έχει κλείσει τα σύνορα με την Ελλάδα με το πρόσχημα ότι δεν θα περάσουν προς τα εκεί πρόσφυγες μετανάστες. Αυτά όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι πράξεις οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία καλών σχέσεων γειτονίας και οπωσδήποτε δεν πρέπει να τις επικροτούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλέκενστάιν, εσείς εισήγητης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ε, λίγες φράσεις μόνο. Τρία, τρία θέματα. Αφενός ότι είπαμε και συμφωνήσαμε ιδίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της δικαιοσύνης ότι θα παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά, να κάνει το λεγόμενο monitoring για να διαπιστώσει ότι όντως προχωρεί η αναθεώρηση του συστήματος της δικαιοσύνης και να δει εάν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε. Σε συνεργασία με τον συνάδελφό μου Κούκαν αύριο θα καταθέσουμε προφορική τροπολογία επί της συμβαστικής τροπολογίας υπαριθμών 6 για να διαγραφούν τρεις λέξεις που αναφέρονται στο αγγλικό enforcement δηλαδή αυτές που λένε and its enforcement και την εφαρμογή της. Δηλαδή αν περιμένουμε όλα αυτά να έχουν εφαρμοστεί τότε γνωρίζουμε ότι αυτό θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Δεν θέλουμε όμως να περιμένουμε τόσο πολύ μέχρι ότου αρχίσουν οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να αποφασιστεί να εγκριθεί στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Θέλουμε να αρχίσει η εφαρμογή implementation started, αλλά να περιμένουμε τώρα μέχρι ότου εφαρμοστούν όλα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δίκαιο και απέναντι στην Αλβανία, διότι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι το έργο αυτό. Να πω μια τελευταία λέξη για αυτά που είπε ο κ. Κούκαν σε σχέση με το νόμο περί μέσων και την πρόσκληση του Γενικού Διευθυντού. Συμφωνώ. Και εγώ θεωρούσα την προηγούμενη νομοθεσία καλύτερη αλλά πρέπει κανείς να δεχθεί κιόλας ότι για πολλά χρόνια ένα μέρος της πολιτικής τάξης στην Αλβανία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να προβάλλει κολλήματα. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να μπορέσει να πληρωθεί η θέση αυτή. Γι' αυτό και εγώ ε, έχω, πώς να πω, είμαι διχασμένος και μέσα μου. Γνωρίζω το ιστορικό, αλλά κάποιος, ε, κάποια λύση πρέπει να βρεθεί ο πρόεδρος. Αύριο θα είναι η ψηφοφορία, είναι. Το μικρόφωνο σας παρακαλούμε. Για Βοσνία γοβίνη τώρα. Ο κύριος Νταν Πρέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες που την προηγούμενη εβδομάδα στήριξαν την ιδέα μετά την ψηφοφορία τον Απρίλιο της έκθεσης για την Βοσνία δηλαδή η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επισκεφθεί τη χώρα. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες. 169 τροπολογίες υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους, όλες τις πολιτικές ομάδες που έδειξαν τέτοιο ενδιαφέρον. Είναι συγκρίσιμο με το τι έγινε και πέρυσι με τις τροπολογίες. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη λοιπόν είναι κάτι που ενδιαφέρει σε συνεχή βάση την Επιτροπή μας. Προσπάθησα λοιπόν να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου όσο γίνεται περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές, τις συμβαστικές τροπολογίες που ετοίμασε. Και έτσι καταλήξαμε σε 19 τροπολογίες που καλύπτουν 115 από τις 169 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. 19 τροπολογίες λοιπόν που καλύπτουν 115 τροπολογίες από τις 169 και αυτό χάρη στην προσπάθεια όλων των πολιτικών ομάδων για να επιτευχθεί συνένεση. Πριν λοιπόν προχωρήσω και μπω στις λεπτομέρειες των συμβαστικών αυτών τροπολογιών, ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές από όλε τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ επίση και τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τη Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο, τον κύριο Πίτσολα, ο οποίος συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μας. Τώρα, πολλές τροπολογίες είχαν να κάνουν με τι πιο πρόσφατες εξελίξεις, με την υποψηφιότητα για προσχώρηση, για τις εξελίξεις του μηχανισμού συντονισμού, για την ε, έγκριση διαπραγματευτικής θέσης όσον αφορά την προσαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθερότητας μετά την προσχώρηση της Κροατίας και συντάξαμε και τις συμβαστικές τροπολογίες 1 και 2 με τις οποίες στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι την ίδια εβδομάδα όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνούσε με τον Κάμερον για την περίφημη προσπάθεια αποφυγής του Brexit, την ίδια εβδομάδα η Βοσνία Ερζεγοβίνη υπέβαλε αίτηση για προσχώρηση. Συμβολικό λοιπόν. Ξεκίνησε η εβδομάδα με αυτήν τη σημαντική χειρονομία της Βοσνίας και ολοκληρώθηκε η εβδομάδα με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τον Κάμερον. Συμβολικά όλα αυτά πολιτικά. Συνεπώς, χαιρετήσαμε την αίτηση για προσχώρηση της Βοσνίας και ζητήσαμε από το Συμβούλιο να εξετάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την υποψηφιότητα αυτή, ώστε να προχωρήσει να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνωμοδότηση. Ξέρουμε ότι η προετοιμασία ε, των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο θα πάρει πολύ χρόνο, οπότε η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει. Η συμβαστική τροπολογία 2 σημειώνει ότι το Συμβούλιο μπορεί να στείλει την υποψιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βοσνία από την πλευρά της πρέπει να προχωρήσει σε δύο κυρίους τομείς, στον ε, συντονιστικό μηχανισμό και στην προσαρμογή του παρικού τμήματος της Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά σημεία. Και αυτά τα δύο σημεία θα βοηθήσουν να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο. Τώρα για μας ο μηχανισμός συντονισμός πρέπει να εναρμονιστεί μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Η διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς να υπάρξει αυτός, αυτή η αλλαγή στο μηχανισμό. Τώρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο για να αποφασίσουμε τι απάντηση θα δώσουμε στο αίτημα προσχώρησης της Βοσνίας. Ο Επίτροπος Χάν είναι στο Σαράγεβο σήμερα για να συζητήσει πάνω σε όλα αυτά τα σημεία. Περιμένουμε επίσης σήμερα και μια λύση για το θέμα αυτό του μηχανισμού συντονισμού, που είναι όπως είπαμε κάτι αναγκαίο. Να υπάρξει εναρμόνιξη μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Θέλω να πω δύο λόγια και για τη συμβαστική τροπολογία 3, η οποία αναφέρεται στην αναγκαιότητα συγχρόνω να συνεχίσουν οι πολιτικέ μεταρρυθμίσει για να γίνει η Βοσνία ένα αποτελεσματικό κράτος που θα λειτουργεί καλά, όπου θα υπάρχει ισότιμη αντιπροσώπευση όλων των πλευρών που συνθέτουν τη χώρα αυτή και να αντιπροσωπεύονται όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως προέλευσης θρησκευτική ή άλλης. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη. Η Κοπεχάγη, το κοινοτικό κεκτημένο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τονίζουμε επίσης την ανάγκη πρόθεση των ευρωπαϊκών αξιών βάσει των αρχών που πενθυμίσαμε και πέρυσι. Φεντεραλισμό, αποκέντρωση και νόμιμη αντιπροσώπευση. Είμαι όμως κάπως απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα συμβασμό όσον αφορά τις εκλογές γενικά και πιο συγκεκριμένα τις τοπικές εκλογές. Επρόκειτο για τις τροπολογίες 68, 109 και 169. Προσωπικά, εγώ δεν έβλεπα προβλήματα όσον αφορά την νόμιμη αντιπροσώπευση όλων των πλευρών και όλων των πολιτών. Ελπίζω μέχρι αύριο η σοσιαλιστική ομάδα να δείξει την αλληλεγγύη που περιμένουμε. Να υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη και εκεί. Γιατί απλώς θέλουμε να επιμείνουμε για το ότι οι εκλογές και κυρίως οι τοπικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη αυτή νόμιμης αντιπροσώπευσης που ζητάνε οι διάφορες κοινότητες στη Βοσνία. Συμβαστική τροπολογία 4 τώρα έρχεται στο δημοψήφισμα στη Ρεπούμπλικα Σπρέσκα. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει. Το δημοψήφισμα αυτό κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τώρα πολλές τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πολύ ευαίσθητο σημείο αυτό με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματο. Κάθε φορά που μιλάμε για διαφθορά, εγώ επιμένω και λέω ότι είναι ένα θέμα πολιτικών κομμάτων πρώτα απ' όλα. Τα πολιτικά κόμματα είναι αυτά που πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουν να εγκαταλείψουν τη διαφθορά. Γιατί η πηγή της διαφθοράς, δυστυχώ βρίσκεται στα πολιτικά κόμματα. Στη συνέχεια, Εντάξει, δεν θα μιλήσω και για τις 19 συμβαστικές τροπολογίες. Έρχομαι στη συμβαστική 11 που αναφέρεται σε σημαντικές ουσιώδεις βελτιώσεις που είναι αναγκαίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τις διακρίσεις σε βάρος μιλάμε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Σόσνη και λέμε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις αυτές. Συμβαστική 16. Εδώ λέμε ότι ανησυχούμε όλου ιδιαίτερω όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και για τα μέσα ενημέρωση και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα και επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης. Η συμβαστική αυτή τροπολογία αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση, πολύ δύσκολη, αφόρητη ε, θα έλεγα, όσων ε, μεταδίδουν εκπομπές. Θα σταματήσω εδώ. Αύριο ελπίζω θα ψηφίσουμε μια δυνατή έκθεση η οποία θα βοηθήσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Κούκαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την έκθεσή του. Η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τα επιτεύγματα της Βοσνίας τους τελευταίους μήνες και αναφέρεται στο τι θα πρέπει να γίνει ακόμα έτσι ώστε να εμπλακεί στην διαδικασία ένταξης. Η πορεία προς εκεί συμβαδίζει με ε, τα βήματα για την βελτίωση της δημοκρατίας στη χώρα, την αναθεώρηση του δικαστικού ε, σώματος, την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε όλα αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Η αποτυχία επίτευξης των στόχων αυτών δυστυχώς δημιουργεί αποκλήσεις από τα standards του ΟΑΣΕ βασικός μας στόχος είναι να ενθαρρύνουμε την Βοσνία ερζεγοβινη να καταστεί μια χώρα η οποία να υποδέχεται με σωστό τρόπο όλους τους πολίτες της και όχι μόνο τμήματα των πολιτών της. Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε επίσης την σημασία που έχει η διακυβερνητική συνεργασία, η διακοινοβουλευτική συγγνώμη, συνεργασία με άλλα κοινοβουλευτικά σώματα και ελπίζω η Κοινή Επιτροπή να υιοθετήσει γρήγορα τους κανόνες λειτουργίας της. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Λέω ο κύριος Καν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την προσπάθεια που έκανε και για το πνεύμα συνεργασίας. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες έχουν γίνει δεκτές η καταπολέμηση της διαφοράς, η καταπολέμηση του αποκλεισμού, παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά, προστασία των μειονοτήτων και των μειονοτήτων των ομοφιλοφίλων. Παρ' όλα αυτά προτείνουμε να υπάρξει μια καταδιέρεση ψήφος το 109 για την πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Η πρότασή μας είναι να αφαιρεθεί η φράση «τρεις συστατικοί λαοί και άλλοι». Η διατύπωση αυτή έχει σχέση με το παράρτημα 4 της Συμφωνίας του Ντέιτον και έχει συμπεριληφθεί και σε άλλο τμήμα της συγκεκριμένη έκθεσης. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του νέου, της πρότασης του νέου εκλογικού νόμου. Το Κοινοβούλιο μας έχει ξεκαθαρίσει ότι περιορισμοί με βάση την εθνότητα ή τον τόπο κατοικίας σε σχέση με την δυνατότητα του εκλέγην και του εκλέγεστε θα πρέπει να μην περιλαμβάνεται στην πρόταση του εκλογικού νόμου σύμφωνα και με την πρόταση του Δικαστηρίου ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με τις προηγούμενες αποφάσεις μας, θα πρέπει να βάλουμε τη φράση όλοι οι πολίτες. Περαιτέρω, θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πραγματικά συνενετική, χαιρετίζει την πρόοδο της Βοσνίας και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Να τελειώσω λέγοντας ότι βασικός στόχος αυτού του Κοινοβουλίου είναι οι εκθέσεις προόδου να είναι απολύτως αντικειμενικές. Πρέπει να προστατεύσουμε την αρχή αυτή εφόσον θέλουμε να θεωρηθούμε αξιόπιστοι εταίροι απέναντι στους ομολόγους μας, όλα δηλαδή τα πολιτικά κόμματα της Βοσνίας Ευζεγοδίνης. Θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε ε, μια ειρηνική εξέλιξη για τη χώρα αυτή με εγγύηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για όλους τους Βοσνίους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάτμανς. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο κύριο Ράντος για την απουσία του και να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Πρέντα για τις 19 συμβιβαστικές του τροπολογίες, δίκαιες και ισορροπημένες τροπολογίες. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή για μια ακόμη φορά να συγχαρώ τη Βοσνία Ευζεγοβίνη για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβεβαιώσω την στήριξή μας στο ευρωπαϊκό μέλλον της Βοσνίας Ευζεγοβίνης η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, όμως η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός συνεργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσλειτουργίες, υπάρχει έμβια και μια πολύ περίπλοκη μορφή εσωτερικής λειτουργίας. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προβλήματα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία ένταξης αφεαυτής είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει εν πολλής για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την ανησυχητική κατάσταση των 85.500 εσωτερικά εντοπισμένων, έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Βοσνία Ευζεγοβίνη και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως επίσης και τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό αγνοουμένων. Εδώ τα βήματα προόδου είναι περιορισμένα. Τα, οι αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν σωστά, να φέρουν σε συνεργασία και τις δύο οντότητες έτσι ώστε να ενισχυθεί η προσπάθειά τους. Ο επόμενος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέντα, εισηγητή, καθώς και τους κύριους εισηγητές, για την συνεργασία και τον διάλογο την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, οι συζητήσεις που διεξαγάγαμε είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα και σημαντικές προκλήσεις. Κατά πολέμηση διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, σημαντικές ελλείψεις ε, στην ελευθερία του τύπου, άσχημη οικονομική κατάσταση στην χώρα που οδήγησε και σε εγκατάλειψή της από πολλούς ε, νέους εγκεφάλους, προβλήματα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι η Υπάρχουν εδώ και κάποιες κινήσεις που γίνονται με πολιτικά κίνητρα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, θέτοντας την έτσι σε ένα άσχημο φως. Ωστόσο δεν θα ήθελα να είναι υπερβολικά αντικέ οι διατυπώσεις. Νομίζω και το εκτιμώ ότι ο εισηγητής έχει στοχεύσει ιδίω στα θετικά. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους πιο δυσίγητες. Η Βοσνία Σεγοβίνη τον Φεβρουάριο κατέθεσε επίσημη αίτηση για ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή, η κατάσταση φαίνεται να καλυτερεύει. Χρειάζεται όμως τη βοήθειά μας η Βοσνία Σεγοβίνη. Έχω να πω και κάτι για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ότι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό μπορέσαμε σε συνεργασία με τους πιο δυσηγητές να καταθέσουμε συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες όμως δεν συμφωνούμε με όλες. Στην τρία όπου απευθύνεται έκκληση για να υπάρξει μια διάκριση σε βάση εθνικών κριτηρίων. Αυτό όμως ε, δεν μπορεί να μα βρει σύμφωνο, διότι έρχεται και αντίθετο στην απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι οι θεσμοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη στην Δημοσιακή να επιλύσουν το πρόβλημα με συνεργασία που θα τους προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η προαναφερθής απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Υφίστανται διακρίσεις ακόμη ένας αριθμός πολιτών. Αυτά τα έχουμε πει κατά επανάληψη και στις συζητήσεις με τους κοιορισίγητες. Και δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή διατύπωση και μια συμβαστική τροπολογία προκειμένου. Πάντως, εάν, δηλαδή να συμφωνήσουμε τη συμβαστική τροπολογία, αν η συμβαστική τροπολογία παραμείνει αύριο, στην ψηφοφορία, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Τώρα, για την τροπολογία 18. Για τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Εμείς χαιρόμαστε για την τροπολογία αυτή. Δεν συμφωνούμε όμως που εδώ τονίζεται μονάχα ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ υπάρχουν πολλά. Ολόκληρη λίστα από περιβαλλοντικά προβλήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Αυτά θα κοιτάξουμε να τα ε, περιλάβουμε στο ε, αντίστοιχο ψήφισμα του χρόνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα, τον εισηγητή και όλους τους σκιώδης. Ευχαριστώ και τον επικεφαλής αντιπροσωπείας για τη σχέση μας με την ε, Βοσνία, τον κύριο Πίτσουλα. Αυτό που είναι ζωτική σημασίας είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει, παρουσιάζει την έκθεσή της όσον αφορά την ε, πρόοδο της χώρας, να έχουμε υπόψη μας ότι το Φεβρουάριο η Βοσνία Ριζεγοβίνη υπέβαλε αίτηση για ένταξη. Η Ολλανδική Προεδρία και το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει τώρα και να επεξεργαστεί το αίτημα αυτό έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 και 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν με άλλες ε, αιτήσει χωρίς καθυστέρηση από το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό λοιπόν κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας το Συμβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται τη γνωμοδότησή της όσον αφορά την αίτηση αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι ένα στοιχείο κλειδί στην διαδικασία αυτή είναι επιπλέον προσπάθειες και κίνητρα προς όλα τα θεσμικά όργανα, όλους τους θεσμούς της Βοσνίας εζεγοβινης ώστε να προχωρήσουν σε παρετέρω μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό πρέπει να σταλούν ερωτηματολόγια. Η διαδικασία διεύρυνσης είναι πολύ απαιτητική ο βαθμός με τον οποίο τα διάφορα όργανα της νετούσης ε, χώρας με στην όλη διαδικασία είναι καθοριστικό. Και στην περίπτωση αυτή επίσης για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ζωτική σημασία μόνο για τους πολίτες της Βοσνίας Ζεγοβίνης, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη της χώρας αυτής. Και αυτό το λέω εξαιτία των αποσχιστικών ε, προσπαθειών. Ακούω ότι ο κύριος Άνοπος και πέρυσι είχε κάποιες ε, επιφυλάξεις Εδώ έχουμε διαφωνήσει επί της αρχής. Άλλη είναι η πραγματικότητα στη χώρα και άλλη είναι η κατάσταση που ορισμένοι θα θέλανε να είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Έτσι κι πρέπει να τηρείτε το Σύνταγμα. Και πρέπει να επιμείνουμε για ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Κυρίως μάλιστα όταν μιλάμε για μελλοντικέ συνταγματικέ μεταρρυθμίσεις. Ο Επίτροπος Χάν λοιπόν πολύ χαίρομαι που βρίσκεται σήμερα στο Σαράγεβο. Συναντιέται με τις αρχές εκεί, κάτι το οποίο σίγουρα θα έχει θετικές επιπτώσεις στην όλη διαδικασία. Θα προωθήσει μια νέα προσέγγιση υπέρ των μεταρρυθμίσεων και επιπλέον ο κύριος Χάντ θα μπορέσει να μιλήσει με τον κύριο Ζιμπέκαβιτς προκειμένου να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να προωθήσουν τον μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα. Θέλω να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στο θέμα της επιστροφής όλων των προσφύγων στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Κυρίως των Κροτών και των Βοσνίων. Ε, έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και χαίρομαι για τις προσπάθειες που έχει κάνει ο κύριος Τσόρτας, αλλά η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει και αυτή να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να, να επιστρέψουν. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική ακόμα η προσπάθεια δηλαδή. Στις ε, μετέπειτα συνεννοήσεις που θα γίνουν μεταξύ των ε, πολιτικών εταίρων και των αρχών ελπίζω να εγκριθεί και ένας νέος εκλογικός νόμος που επίση είναι ζωτική σημασία για να μπορεί να λειτουργεί καλά η χώρα. Ελπίζω ότι στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρεθεί μια λύση τελικά. Και αυτό για να προχωρά και απρόσκοπτα η Συμφωνία Σταθερότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια διαπραγματευόμαστε πάντως και στο μέλλον όλοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η Βοσνία και η Ριζακοβίνη να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Hvala gospodine predsjedniče. Nakon kruga pregovora pohvalio bi napor izvjestitelja gospodina. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα προσεκτικά τον πρώτο γύρο των συζητήσεων και θέλω να συγχαρώ επίσης και τον κύριο Πρέντα για μια αντικειμενική παρουσίαση για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο προηγούμενος χρόνος ήταν ένας θετικός χρόνος για τη συγκεκριμένη χώρα. Όλοι οι ηγέτες, οι πολιτικοί της Βοσνίας Ζεγοδίνης υπέγραψαν την συμφωνία αυτή για τις μεταρρυθμίσεις. μετά από την η κατάθεση της αίτηση για την ένταξη της χώρας. Η Βοσνία Ευζεγοβίνη πλέον έχει καταθέσει την αίτησή της για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται προσπάθειες για να βγει κανείς από το αδιέξοδο του πλαισίου Dayton. Όλοι θα πρέπει να στηρίξουμε την συγκεκριμένη αυτή αίτηση. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος Χαν θα επιτύχει στις διαπραγματεύσεις του με τους ηγέτες τους πολιτικούς της χώρας. Ιδιαίτερα στον τομέα της εφαρμογής και της Συμφωνίας Συνεργασίας αλλά και των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν Πάντα περιμένουμε να γίνει απογραφή πληθυσμού. Δεν έχουν υπάρξει βήματα προόδου από πλευρά της κρατικής μηχανής και αυτό δεν επιτρέπει στην χώρα να προχωρήσει στην δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών. Υπάρχουν λοιπόν συστημικά προβλήματα, θα πρέπει οι καταγγέλλοντες σαν παράδειγμα να προστατεύονται και το θέμα της ε, μεταρρύθμισης της δικαστικής εξουσίας είναι κάτι στο οποίο απαραίτητα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έτσι ώστε η Βοσνία Ευζεγοβίνη να γίνει μια χώρα λειτουργούσα βασισμένη στην επικουρικότητα, την ισότητα ε, όλων των συνιστοσών των εθνοτικών. Λυπάμαι λοιπόν γιατί μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα κοινό σώμα συνεργασίας ανάμεσα στην Βοσνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε τις προβλέψεις του Dayton, οι οποίες προβλέπουν οι απογραφές να γίνονται σε εθνοτική βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ένα σύντομο σχόλιο υποστηρίζοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καν. Εκπροσωπεί την πολιτική μας ομάδα συνολικά όταν αναφέρεται σε σχέση με τον όρο ε, εθνοτικές συνιστώσεις η δική μου πολιτική ομάδα προσπάθησε να βρει μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Από τη μία θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε το σεβασμό του Dayton, των προβλέψεων του Dayton. Από την άλλη θέλουμε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός έτσι ώστε η Βοσνία να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην μείνει μόνο με τις προβλέψεις του Dayton. Πέρυσι ε, κάναμε προσπάθειες ε, σαν πολιτική ομάδα και καταφέρουμε να μην αναφερθούμε στους λαούς που συνιστούν τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά συνολικά στη χώρα αυτή. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο κύριος Καν είναι να υπάρξει η αναφορά αυτή στην έκθεση έτσι ώστε να δείξουμε ότι θέλουμε να υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε επανειλημμένα την αναφορά αυτή και να περιοριστούμε στην άπαξ αναφορά της έκφρασης. Λοιπόν, η ομάδα μας έχει αλλάξει την αρχική της θέση, αναζητεί ένα συμβιβασμό και δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε χώρο για πολιτικές διαφορές. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ουσιαστικό συμβιβασμό γιατί ουσιαστικά εμείς λέμε ε, στους Βοσνίους να βρουν ένα συμβιβασμό και πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα για να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ. ερμήνευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αίτηση της Βοσνίας ε, σαν μια ξεκάθαρη επιθυμία να περάσουν από τον Dayton στις Βρυξέλλες, να μειωθεί το εθνικό δηλαδή χαρακτηριστικό και να αυξηθεί η ιδιότητα του πολίτη στην συνταγματική τάξη της χώρας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μπλοκαρίσματος που συνοδεύουν τον χαρακτηρισμό της χώρας σαν μια χώρα που αποτελείται από τρεις εθνοτικές συνιστώσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί όταν ε, γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία. Λοιπόν, η επιμονή στους όρους στους οποίους αναφέρθηκε και ο τελευταίος ομιλητής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η Βοσνία σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο πάλι. Άκουσα το όνομα Σαφχάουζερ και φοβήθηκα, λέει ο κύριος Πρέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας. Έχει γίνει αρκετή προσπάθεια μέχρι τώρα και αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι το εξή. Είδατε ότι πέρυσι όλοι συμφώνησαν έτσι ώστε να παραμερίσουμε λίγο την συζήτηση για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να συγκεντρώσουμε την προσοχή στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτείται να γίνουν στον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι σοσιαλιστές. Και τελικά η διαφωνία μας γίνεται στα πλαίσια της αναφοράς του όρου ε, συστατική λαή, συνιστώντες λαή. Αυτό είναι κάτι που άπτεται της ε, θεσμικής αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης χώρας. Υπάρχει ανάγκη και αυτό έχει αναγνωριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να υπάρξει πρόοδος βέβαια στα συνταγματικά και θεσμικά προβλήματα. Εγώ διαπιστώνω ότι οι σοσιαλιστές πράγματι ε, μετακινήθησαν λίγο και πράγματι θέλουν να υπάρξει αναφορά στον όρο αυτό έστω και μία φορά. Οπότε θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα το επιχείρημα του κυρίου Χάουιτ θα πω δηλαδή ότι ε, πράγματι σε ένα έγγραφο αρκεί να υπάρξει μία συγκεκριμένη αναφορά ενός όρου και σε άλλα θέματα. Γιατί στο 99% των περιπτώσεων οι σοσιαλιστές επιμένουν να εγγραφεί σε όλο το κείμενο ακριβώς η ίδια αναφορά. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ξεχάσω την πρότασή τους, θα πρέπει όμως να αποφασίσουμε μέσω ψηφοφορίας ε, το θέμα της αναφοράς στους λαούς, τους επιμέρους της χώρας, ιδιαίτερα σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ότι δυστυχώς όλη η προσπάθεια η οποία έχει γίνει έχει μπλοκαριστεί από αυτό το οποίο είπε ο κ. Πιτσόλα δηλαδή το θέμα της, ε, ε, της καταμέτρησης του πληθυσμού, της απογραφής. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και τα δεδομένα, τα καταγραφικά τα οποία έχουμε είναι δυστυχώς αμφισβητούμενα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την συγκεκριμένη χώρα αν προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι η αναφορά στο συνταγματικό πλαίσιο είναι δευτερεύουσα και ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια ερμηνεία του συντάγματος της Βοσνίας της Ζεγοδίνης σεβόμενοι ορισμένες πλευρές χωρίς να μπούμε όμως σε μια αυστηρά νομική ανάγνωση. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο παραπέμπει στην εθνή εθνοτικοποίηση της πολιτικής δραστηριότητας. Αυτή η δισκαμψία των θέσεων ορισμένων πολιτικών ομάδων, την οποία εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Δεν ξέρω γιατί η αναφορά στους συστατικούς λαούς παραπέμπει σε μια εθνοτικοποίηση της πολιτικής δραστηριότητας στη χώρα και δεν ξέρω ε, αν, πώς θα παρεμποδίσουμε τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα αν αποκρύψουμε την αλήθεια. Συνεπώς λοιπόν εγώ περιμένω με ανυπομονησία την ψηφοφορία αύριο και για μια ακόμη φορά είμαι ευγνώμων στους φίλους όλων των πολιτικών ομάδων για την προσπάθεια την οποία έκαναν με στόχο να επιτευχθεί συγκεκριμένη συμβιβαστική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ήταν θυμίζω 115 οι τροπολογίες οι οποίες συνοψίστηκαν σε συμβιβαστικές. Ο κύριος Πρέγκοβιτς ζήτησε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχόλιο για το θέμα που δεν είναι βεβαίω τεχνικό, είναι εξόχως πολιτικό και συμφωνώ με τον εισηγητή κύριο Πρέντα. Ωστόσο, μια αναφορά στα όσα είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Βεβαίως και εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε τη Βοζήρα Ζεγοβίνη από τον Τέιτον στις Βρυξέλλες. Και μάλιστα ίσως να εργάζομαι το ίδιο σκληρά και εγώ καθημερινά όσο και εσείς. Θα προτιμούσα να μας είχατε πει λίγο περισσότερο για τα βασικά μηνύματα του Επιτρόπου Χάν σήμερα στο Σαράγεβο. Αντί να μιλήσετε δικά κάτι σαν να είναι ξεπερασμένο. Όχι, αντίθετα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέρος του συντάγματος. Δεύτερο, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος εάν σας χορηγήσει το Συμβούλιο εντολή αρχίσετε να προετοιμάζεστε ο Επίτροπος σας φάνηκε πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για την προετοιμασία της πορείας της Ορθέδης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε πολύ διότι δεν ήταν διόλου προφανές αυτό ως εξέλιξη. Αναμένουμε λοιπόν και επιθυμούμε να δούμε την Κομισιόν να εργαστεί για την πορεία της χώρας αυτής από τον Τέιτον μέχρι τις Βρυξέλλες αλλά για να, πράγμα, ε, ε, δικαιωθούν και οι ελπίδες του λαού αυτού. Σας ευχαριστώ. Το Dayton αρκούσε ίσως για να λήξει τότε ο πόλεμος. Δεν αρκεί για να εξασφαλίσει το μέλλον της χώρας αυτής. Χρειάζεται ένα ποιοτικό άλμα και το ποιοτικό άλμα αυτό άλμα για να γίνει χρειάζεται εξωτερική βοήθεια αλλά χρειάζεται και εσωτερικές διαδικασίες. Η δεμή δεν βλέπω και πολύ μεγάλες πιθανότητες σε ό,τι αφορά μια πρόοδο προς την ένταξη. Για μένα αυτό είναι πολύ ξεκαθαρό. Ότι δηλαδή εναπόκειται και στις προσπάθειες των ίδιων των Βοσνίων και δεν θα έπρεπε να γύρονται ελπίδες οι οποίες δεν είναι δικαιολογημένες. εάν δεν έχουν επιληθεί δηλαδή αυτά τα πολύ ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε ήδη δεχτεί στους κόρπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές, επιβολικά πολλές χώρες όπου δεν καταφέρνουμε να λύσουμε τα προβλήματά τους ούτε εκ των υστέρων. Αυτά πρέπει να λεχθούν ξεκάθαρα. Και μια ενδιάμεση παρατήρηση. Μόλις διάβασα μια είδηση από τη ρωσική εφημερίδα Ισβέστια πρώην της ρωσικής κυβερνήσεως ίσως και σήμερα ακόμα που λέει ότι τον Απρίλη θα μεταβεί ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε οικονομική διάσκεψη στην Κρυμαία. Για μένα είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως πρόκειται για μεμονωμένους ευρωβουλευτές, αλλά δεν μπορούν αυτοί να θεωρηθούν ούτε να θεωρήσουν ότι είναι ότι αντιπροσωπεύουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει να διασαφηθεί και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα, υπαριθμόν 6. μελλοντική καινοτόμως στρατηγική για το εμπόριο και τας επενδύσεις. Νέα, μακρόπνοη και καινοτόμος. Δεν έχω δει ποτέ καμία ε, καινοτόμο αλλά όχι νέα. Δεν θα είχε λογική κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο τίτλος μου φαίνεται λίγο παράξενος. Τα Σάφη είναι η συγκεκριμένη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, γενικά μιλώντας η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και συνεισφέρει στην πρόθεση των αξιών της. Εξάλλου έχει χρησιμοποιηθεί στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του εμπορίου που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Είμαι συγγήτρια για τη συντάκτρια μάλλον της νομοδότησης αυτής που αναφέρεται στην ε, εμπορική πολιτική της Ένωσης στο μέλλον. Εγώ θέλησα να επικεντρωθώ στο διεθνές εμπόριο από πλευρά των εξωτερικών υποθέσεων και στα πλαίσια των ε, διεθνών σχέσεων. Κάθε παράγραφος λοιπόν αντιστοιχεί σε μια κεντρική ιδέα. Πρόκειται καταρχήν για το εξή. Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εμπορική της πολιτική, η οποία πρέπει να σέβεται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θέλησα να επιμείνω στη σημασία που έχει η εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών και κυρίως όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη που προστατεύει και το περιβάλλον. Και θέλεις επίσης να υπενθυμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει ο καλός συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους παίκτες της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της διαφάνειας. 65 τροπολογίες υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης και εμείς καταλήξαμε σε 14 συμβαστικές τροπολογίες που περιλαμβάνουν τις περισσότερες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και τις ιδέες τους. Ελπίζω λοιπόν ότι θα τις στηρίξουν οι πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους και όδες εισηγητές για την καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας και περιμένω τις παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος, δεν τον ακούμε. Grazie, sostituisco il collega. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Μπενιφέη, ο οποίο ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Να ευχαριστήσω την κυρία Σεφή. Είναι ένα καλό κείμενο, ένα ισορροπημένο κείμενο αυτό το οποίο προτείνει. Οι αναφορές που γίνεται που γίνονται ε, στις εξωτερικές εμπορικές δραστηριότητες σαν διπλωματικό μέσο και σαν χρήσιμο μέσο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αηφόρου ανάπτυξης. Έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις της εμπορικές όλο ένα και πλέον διαφανείς και προσβάσιμες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς καταθέσαμε τροπολογίες για να υπογραμμίσουμε περαιτέρω συγκεκριμένα σημεία τρία θέματα. Ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και διεθνές υπολιμερές πλαίσιο. Ε, μαζί με τις αρχές του καθολικού και του αδιέρετου χαρακτήρα των δικαιωμάτων υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο για την συμπερίληψη δεσμευτικών ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα εργασιακά δικαιώματα υπενθυμίζουμε τον κεντρικό χαρακτήρα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων, της συνεργασίας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού όλων αυτών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογραμμίσαμε επίσης και την πολυμερή διάσταση, την σημασία που έχει η συνοχή στην εξωτερική μας εμπορική πολιτική και στα πλαίσια της ε, ανάπτυξης μέχρι το 2030 και να γίνει αναφορά στη συμφωνία την οποία καταλήξαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο για την προσαρμογή στη σημερινή οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει όλες οι προτάσεις μας περιλαμβάνονται στις τροπολογίες που καταθέσαμε. Ευχαριστώ την κυρία Σαϊφή για το επικοδομητικό πνεύμα το οποίο επέδειξε. Γιατί έτσι βελτιώνεται ένα κείμενο το οποίο έτσι κι αλλιώς εξ αρχής ήταν ένα καλό κείμενο. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες και δει την υπαριθμόν 13 εξαγωγές όπλων εξοπλισμού. Παλαιά επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εξαγωγές εξοπλισμού να ρυθμιστούν δεσμευτικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταργηθούν οι σχετικοί περιορισμοί. Αυτός ο κώδικας διοντολογίας, Code of Conduct, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει δεσμευτικό. Να μπει αυτό στην 13 και να ζητήσουμε ότι ο Code of Conduct για τις εξαγωγές εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει δεσμευτικό. Ίσως εσείς κυρία Συγήτρια μπορείτε να το περιλάβετε στις συμβαστικές αστροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν επιθυμεί άλλος να λάβει το λόγο. Η κυρία Σαϊφή. Εντάχει κύριε Πρόεδρε, για αυτό που μου ζητήσατε θα το εξετάσω. Είναι βέβαια κάπως περίπλοκο το θέμα. Θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Παντζέρη. Συνεργαστήκαμε όντως πολύ επικοδομητικά για τον φάκελο αυτό και πολλά θέματα που ζήτησαν οι συνάδελφοι των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, ενσωματώθηκαν στο εγγραφό μου. Αυτά σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη η συνεδρίαση. Αύριο το πρωί.